Καλημέρα σε όλους. Ξεκινάμε την συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Είναι ιδιαίτερο πλούσια στην ημερήσια διάταξη. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, ε, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Η σημερινή συνεδρίαση αναμεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Ξεκινάμε με το σημείο 3, αλλά πρώτα θα ήθελα να χαιρετήσω μια πολύ αριθμή αντιπροσωπία των μελών ε, της Επιτροπής Γεωργίας ε, του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Σήμερα θα ψηφίσουμε και το πακέτο του James Nicholson για το γάλα. Λοιπόν, θα, έχετε, ε, θα, έχει, θα έχει περιεχόμενο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σημείο 3. Κατάργηση ορισμένων παροχημένων πράξεων του Συμβουλίου στον τομέα κοινή γεωργικής πολιτικής. Και εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο τη ε, βελτίωση της νομοθεσίας και έχει ως στόχο τη μείωση των νομοθετικών πράξεων. Έτσι λοιπόν εμείς ε, καταργήσαμε ορισμένες πράξεις μέσα από την κωδικοποίηση ή την προσαρμογή των παλιών πράξεων. Αυτό το σημείο βρίσκεται καθαρά πληροφοριακά στην ημερήσια διάταξη γιατί στάλθηκε η έκθεση στις 3 Ιουνίου το 2011 και επειδή δεν είχαμε αντιρρήσεις ε, μέσα στις 21 ημέρες από την αποστολή του σχεδίου βάσει του άρθρου 46 παράγραφος 2 θεωρείται αυτόματα εγκεκριμένη. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν θέλει να προσθέσει τίποτα. Οπότε πάμε στο σημείο 4. Ειδικά μέτρα στον τομέα της Γεωργίας για τις άκρος απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης. Ο Μάτο Αντροβέρη είναι ο εισηγητής. Εδώ προβλέπει ο σχετικός ε, κανονισμός, ειδικά μέτρα στον τομέα της ε, γεωργίας για τις απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης και που τροποποιήθηκε μετά από την έγκρισή του της 30 Ιανουαρίου του 2006. Η Κομισιόν θέλει να τον τροποποιήσουμε και να τον ευθυγραμμίσουμε και με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θέλει λοιπόν να <coughs> αναδιαρθρώσουμε η Κομισιόν το νομοθετικό κείμενο για να το προσαρμόσουμε στο κάθεστος ε, ΠΟΣΕΙ στο στην ε, Γεωργία. Ο Μάτο, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ΠΟΣΕΙ είναι ένα πρόγραμμα που όπως όλοι γνωρίζετε αφορά στις υπερ ε, περιφερειακές περιοχές της Ισπανίας, της Πορτογαλίας ε, και της Γαλλίας. Εγώ επαναλαμβάνω ότι αν δεν υπήρχε το ΠΟΣΕΙ δεν θα υπήρχε και γεωργία σε αυτές τις απόκεντρες περιφερειακές περιοχές. Για μια ιστορική αναφορά. Αυτό το πρόγραμμα ΠΟΣΕΙ για τις νησιωτικές ε, περιοχές ε, και τις υπερπόντιες περιοχές άρχισε να ισχύει το 81 και σήμερα εννέα περιφέρειες ε, είναι δικιούχοι αυτού του μέτρου. Αυτά τα προγράμματα παίζουν αδιάρρηκτο ρόλο στην διατήρηση της γεωργίας και στην ανάπτυξή τους, όπως επίσης και στη μεταποιητική βιομηχανία αυτών των περιοχών. Και αυτό και λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιφέρειες ε, λόγω της απόστασης από τη Μητρόπολη αλλά και από το μικρό περιθώριο το οποίο διαθέτουν για τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους. Το ΠΟΣΕΗ έχει δύο διαφορετικά καθεστώτα μεταξύ τους. Το ένα αφορά στην αυτάρκεια, δηλαδή να καλύπτονται οι ανάγκες της ε, περιφέρειας αυτής ε, με ε, κοπάδια και με μεταπητική βιομηχανία και γεωργία και μετά είναι το δεύτερο σκέλος που αφορά στην συντήρηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στη διατήρησή τους και την αηφορία τους. Είχαμε πρώτη μεταρρύθμιση το 2001 και η δεύτερη, την πιο σημαντική, το 2006, όπου έγινε και μία στροφή ως προς την ανάπτυξη των προγραμμάτων που περνάνε στα χέρια της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε μια τέτοια φάση κρίσης ε, οι υπερπεριφερειακές περιοχές υποφέρουν από πολύ ψηλότερα ε, ποσοστά ανεργίας. Πρέπει λοιπόν εμείς να ενισχύσουμε ιδιαίτερα το πρόγραμμα ΠΟΣΕΙ. Όπως είπε ο πρόεδρος στην αρχή, πρέπει να το προσαρμόσουμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ως νομική βάση στο άρθρο 349 της ε, συνθήκης της Λισαβόνας πρόκειται για ένα άρθρο το οποίο εγγυάται διαφορετική μεταχείριση στις άκρως απόκεντρες περιοχές. Και μετά έχουμε και τις ε, βασικές αλλαγές. Μετά βέβαια και στη συζήτηση μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε τα ζητήματα επιτροπολογίας και τα τεχνικά προβλήματα που αφορούν στα προγράμματα. Το ένα είναι το τι στοιχηματίζουμε για την ποιότητα, για τα προϊόντα ποιότητας και ταυτόχρονα θέλουμε να έχουμε και τη χρήση του γραφικού συμβόλου της περιφέρειας αυτής από την οποία προ... της περιφέρειας ε, από όπου θα προέρχονται και τα προϊόντα με ναι, ονομασίες προέλευσης ε, και γεωγραφικής προέλευσης. Πρέπει όμως να εντείνουμε τους ε, φυτοφαρμακευτικούς ελεγχούς, να εξαλείψουμε νοσογο, τους νοσογόνους ε, οργανισμούς, να τους ελέγξουμε και αυτό προωθώντας τα, ε, τους ελέγχους σε όλες ε, τις περιφέρειες. Πρέπει επίσης να ασχοληθούμε με τις γεωργικές ασφαλίσεις για να θα πρέπει να δίνονται ενισχύσεις ούτως ώστε οι ε, επιχειρήσεις, οι γεωργικές επιχειρήσεις να μπορούν να συνάπτουν γεωργική ασφάλιση όπως μας το ζήτησαν και η Επιτροπή Ρέντγι και η Επιτροπή Ίντα. Πρόκειται για μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει να συμβιώσουμε. δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπογράφει συμφωνίες με τρίτες χώρες. Έχουμε τη συμφωνία με την Κολομβία, με το Περού και τώρα υποδιαπραγμάτευση τη συμφωνία με το Μερκοσούρ. Πρέπει όμως να ε, ξεκαθαρίσουμε ότι την τιμή αυτό, το τίμημα αυτών των συμφωνιών δεν θα πρέπει να το πληρώσει η Γεωργία. Θα πρέπει να γίνουν μελέτες επιπτώσεων ούτως ώστε είναι, να διαπιστώνεται αν οι νέε συμφωνίες έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την γεωργία, σε ποιον τομέα και να μπορούμε να βλέπουμε ποιες θα είναι και οι αντισταθμίσεις που θα παρέχουμε. Τώρα, για τις ενισχύσεις στους τοπικούς ε, παραγωγούς ε, τις, ε, ε, τις κρατικές ενισχύσεις με τις ευρωπαϊκές. Θα πρέπει θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα τα οποία δέχονται αυτές τις ενισχύσεις ε, καλύπτουν, όλα τα ζητούμενα, κυρίως στον υγειονομικό τομέα. Και θα πρέπει να δούμε πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις μας σε περιφερειακό επίπεδο. Διότι Κάθε φορά αλλάζουν οι δικαιούχοι. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι το ΠΟΣΕΙ θα περιφρουρεί τις τοπικές καλλιέργειες και θα ευεργετεί τους γιοργούς. Θα πρέπει να δίνονται προκαταβολές στις τοπικές παραγωγές και να λαμβάνονται και άλλα σημαντικά μέτρα. Υπάρχουν βεβαίως οικονομικά μέτρα που όλοι τα περιμένανε και προτείνονται άλλαγες αλλά πρέπει να είναι δικαιολογημένες. Έχει αποδειχθεί ότι είναι ανεπαρκής η πρικοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Υπάρχει οπισθοχώρηση στον τομέα της γεωργίας και χρειάστηκε να υπάρξει και κρατική παρέμβαση για την ενίσχυση της Γεωργίας. 46 εκατομμύρια στην περίπτωση της Ισπανίας, 40 στη Γαλλία για την ντομάτα κλπ. Επίσης η μείωση των δασμών για την εισαγωγή της μπανάνας στις συμφωνίες που υπογράψαμε με την Κολομβία και το Περού προϋποθέτει και μία ενίσχυση στους παραγωγούς. ...30 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την έκθεση η οποία στάλθηκε από την Ίντα για την μπανάνα. Τα οπορικητευτικά, το κρασί, επίσης χρειάζονται αύξηση. Επίσης, λέω ότι οι ελάχιστες εναλλακτικές λύσεις που έχουν τα νησιά και οι απόκεντρες περιφέρειες στην Γεωργία οδηγούν στην ενίσχυση των μέτρων του ΠΟΣΕΗ και αναγνώριση του ποιοτικού άλματος των τελευταίων ετών. Και κάτι άλλο που είναι και προσωπικό θα έλεγα. Θα μπορέσετε να διαπιστώσετε του λόγου του αληθές ε, στην επίσκεψη που θα κάνει αυτή η Επιτροπή στις 31 Αυγούστου στα Κανάρια νησιά. Θα διαπιστώσετε ότι η γεωργία στα, στα Κανάρια νησιά είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι ούτε ενισχύσεις, ούτε μέτρα, ούτε διατάξεις. Είναι περιβάλλον, είναι ομορφιά. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου των τελευταίων μηνών, όπως επίσης και τους ε, συντάκτες νομοδότησης στη Ρέγκη και την Ίντα και πιο συγκεκριμένα στους συναδέλφους από τις απόκεντρες ε, περιφερειακές περιοχές με τους οποίους έχουμε καταπληκτική σχέση και συνεργαστήκαμε πολύ στενά. Τώρα θα ήθελα μέσα από τις τροπολογίες ε, να συνεισφέρετε όλοι και να υποστηρίξετε την έκθεση αυτή που είναι σημαντικότατη για μία περιφέρεια την οποία θα επισκεφθείτε λίγαν συντόμως και θα διαπιστώσετε του λόγου του αληθές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάτο. Ξεκινάει η συζήτηση. Ραντς Γκαρσία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα όχι τόσο να κάνω ερώτηση στον κύριο Μάτο αλλά ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρευρίσκεται. Γιατί ένα από τα σημαντικότερα θέματα που διακυβεύεται εδώ, κυρίως για τη χώρα μου, είναι συγκεκριμένες καλλιέργειες και η κατάστασή τους. Προκειμένου η μπανάνα στα Κανάρια νησιά. Οι Ευρωπαίοι μπάνανοπαραγωγοί έχουν ε, καταθέσει μια μελέτη πρόσφατα και την έστειλαν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επειδή η Κομισιόν σήμερα παρευρίσκεται, όπως είπαμε, θέλω να τη ρωτήσω αν είχε την ευκαιρία να μελετήσει το έγγραφο αυτό και τι ε, γνώμη έχει, τι φρονεί από αυτού, γιατί η κατάσταση είναι πολύ ενισχυτική της μπανάνας στα Κανάρια. Και σε αυτή την έκθεση για το είναι ενδιαφέρον να μάθουμε τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ραντς Γκαρσία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον συνάδελφο Γκαμπριέλ Μάτο για την έκθεσή του, κυρίως διότι ουσιαστικά ο στόχος της έκθεσης ε, δεν ε, ήταν πολύ φιλόδοξος. Θα αναφέρονταν κάποια μέτρα, αλλά θα περιγραφόταν κυρίως στο εφιστάμενο πρόγραμμα POSEI ε, και θα διευκρινίζονταν οι τροποποιήσει που επιφέρει η συνθήκη της Λεσσαβόνας. Αλλά δεν περιορίστηκε σε αυτό η έκθεση. Εγώ ε, ε, έρχομαι από μια περιοχή όπου το 1974 με την Επανάσταση η Γεωργία ήταν σε μια μεσαία μέτρια κατάσταση και με τις δημοκρατικές δυνάμεις και την αυτονομία και την προσχώρηση στην ΕΟΚ το 1985 τότε και με τα προγράμματα μεταγενέστερα από ΖΕΗ το 92 για τις Αζόρες. Χάρη σε όλα αυτά, κατέστησαν δύνατες οι προσαρμογές ε, ε, των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που πρέπει να εξειδικευθούν για περιοχές που απέχουν 2.000 χιλιόμετρα και πάνω από το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κινούνται σε μία σκάλα, σε μία κλίμακα πολύ μικρότερη σε σχέση με το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα δεν πρόκειται μόνο για τη δική μας την περιοχή, αλλά και για άλλες ε, άκρος απόκεντρες ε, περιοχές ε, παρατηρείται μία πολύ θετική εξέλιξη, μία ποιοτική παραγωγή. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε τους περιορισμούς, τα προβλήματα που έχουμε λόγω της κλίμακας της οικονομίας και της απόστασης. Άρα παρόλα αυτά αναπτύσσονται οι τομείς συγκεκριμένα στην περιοχή μου ο γαλακτοκομικό ε, τομέας ε, αντιστοιχεί σε πάνω από 30% της γεωργικής μα παραγωγή. Αυτό κατέστη δυνατό ακριβώς χάρη σε αυτήν την προσαρμογή. Και εξού και το κουράγιο και η τόλμη του Γκαμπριέλ μέσα σε αυτή την έκθεση ζητάει μεγαλύτερη ευελιξία. Ζητάει προσαρμογή των προγραμμάτων ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών για τις μπανάνες παραδείγματος χάρη και είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε τον αντίκτυπο και να θεσπίσουμε κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε να καλύψουμε αυτές τις συνέπειες, ούτως ώστε να μην πληγεί η γεωργία σε αυτές τις περιοχές. Ε, μελλοντικά η ενδεχόμενη κατάργηση των ποσοστώσεων ε, στο γαλακτοκομικό τομέα για τις αζόρες, συγγνώμη, ε, υπάρχει... Ε, ε, η επιτακτική ανάγκη να γίνει αξιολόγηση αντικτύπου, ούτω ώστε τα μέτρα που θα θεσπιστούν να καλύψουν το μελλοντικό ε, σενάριο ε, ανάπτυξη τη γεωργία σε αυτέ τι περιοχέ. Επίση, υπάρχει το θέμα των νέων δυναμικών εξελίξεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση αντικτύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτο ανεφοδιασμού χρειάζονται νέα μέτρα. Κοιτάξτε, θα, όντως ε, θα πρέπει να, ε, τα μέτρα που θεσπίζουμε να αντιστοιχούν στα κονδύλια που έχουμε. Και όταν ζητούμε όμως ευελιξία και νέα δυναμική, είναι επιτακτική επίση η ανάγκη να θεσπιστούν νέα μέτρα, ουσιαστικά μέτρα. Και γι' αυτό σα λέω ότι ο εισηγητή ε, υπερβαίνει αυτό το 20% που προτείνεται ε, για το ειδικό καθεστώ ανεφοδιασμού και τοποθετεί το ποσοστό σε 10% για όλα τα προγράμματα, ούτω ώστε αυτέ οι οικονομίε ε, να προσαρμοστούν γιατί αντιμετωπίζουν ειδικέ δυσχέρειε. Αυτέ οι περιοχέ επίση θίγονται πάρα πολύ από τι φυσικέ καταστροφέ και από τι κλιματικέ αλλαγέ γιατί είναι μέσα στη μέση του ωκεανού Άρα χρειάζονται εγγύσει για να αφοσιωθεί κάποιο ε, στην γεωργία λόγω του κινδύνου των φυσικών καταστροφών. Ε, διότι ο κίνδυνο είναι υπερβολικά υψηλό και μέσα στην έκθεση βλέπουμε την δυνατότητα ad hoc επιδοτήσεων ακριβώ ώστε να είναι δυνατή η συγχρηματοδότηση των γεωργικών εγγύσεων με τρόπο ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο γεωργικέ δραστηριότητε σε αυτέ τι περιοχέ λαμβάνοντα υπόψη την ε, μεγάλη σημασία αυτών των περιοχών και θα κλείσω εδώ πρόεδρε όπως ε, άρχισα ε, ευχαριστώντας δηλαδή τον εισηγητή, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτής της γνωμοδότησης που είναι πολύ πιο φιλόδοξη όπως έλεγα σε σχέση με τον αρχικό στόχο της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μισελ Νταντένι και κατόπιν Μάγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας ε, για την ποιότητα της δουλειάς τους. Οι υπερπεριφερειακές περιοχές πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Είναι, είναι μακριά. Και από το βλέμμα μας και από την καρδιά μας. Είναι τα πρώτα θύματα ορισμένων συμφωνιών που έχουμε υπογράψει με χώρες οι οποίες βεβαίως και χρειάζονται να αναπτυχθούν, αλλά οι οποίες ε, έχουν παραγωγές, οι οποίες ανταγωνίζονται τις δικές μας ε, παραγωγές. Μιλάμε για την μπανάνα, αλλά υπάρχουν ε, προβλήματα όμως και στην παραγωγή του, του ρουμιού. Διότι ανάλογα και με τα οικονομικά δίκτυα ε, καλύπτεται η παραγωγή του Ρωμιού ακόμη και σε αμερικάνικες επικράτειες. Και πέρα από την επίσκεψη που θα έχουμε σε μερικές εβδομάδες σε μία από αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές, θα ήταν καλό στην Επιτροπή μας να έχουμε μία κρόαση για να συζητήσουμε την αντιπροσώπευση αυτών των απομακρυσμένων περιοχών. Α, ξέχασα τον, ε, την Πατραονέδες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Καμπριέλ Μάτο πρώτα απ' όλα. Όχι μόνο μας παρουσίασε μια εξαιρετικά σχολαστική δουλειά που έκανε για τα προγράμματα ε, καλύπτοντας όλες τις άκρες από τρεις περιοχές, αλλά πέραν από αυτό συνεργάστηκε με όλους τους βουλευτές που έρχονται από τις άκρες από κεντρές περιοχές. Ε, συνεργάστηκε στενά και γι' αυτό η γνωμοδότηση αυτή συνιστά μεγάλο άνοιγμα προ όλε τι προτάσει ε, που έχουν γίνει από του βουλευτέ του Κοινοβουλίου και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω. Έχει ζωτική σημασία το ΠΟΖΕ για τη Γεωργία στις ε, άκρως απόκεντρες περιοχές, αλλά έχει και ζωτική σημασία για θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση, με την οικονομία, την οικονομική δραστηριότητα των νησιών, τη γεωγραφική θέση των νησιών και άρα το ΠΟΖΕΙ δεν πρέπει να το εξετάζουμε μόνο σε συνάρτηση με τη γεωργία. Πρέπει να θεωρηθεί ως ένα σφαιρικό συνολικό εργαλείο ανάπτυξη των αρχιπελάγων αυτών των από κέντρων περιοχών της Ένωσης. Ε, προσυπογράφω ε, όλες τις δηλώσεις ε, του Γκαμπριέλ σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα των νησιών και θα ήθελα μόνο να προσθέσω το εξή. Σήμερα αντιμετωπίζουμε μια σοβαρότατη πρόκληση με τις διάφορες διμερείς συμφωνίε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το Μερκοσούρ. Θα ήθελα να τονίσω εδώ, να καταδείξω εδώ ότι τα αποτελέσματα της μελέτης αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Μερκοσούρ, ο αντίκτυπος που θα υπάρχει για τη Γεωργία λοιπόν έχει ως εξή. Οι πλέον ευπαθείς περιοχές, δηλαδή οι άκρος κέντρες περιοχές και οι τομείς, οι ευπαθείς τομείς όπως η παραγωγή ε, του κρέατος ε, στις Αζόρες ε, θα πληγούν όλος ιδιαίτερος και ο αρνητικός αντίκτυπος επί της γεωργίας που θα προκύπτει από αυτή τη συμφωνία θα επιδεινώθει στην περίπτωση αυτών των απόκεντρων περιοχών. Είναι δυσμενέστερη η θέση λοιπόν των άκρος απόκεντρων περιοχών βάσει της συμφωνίας αυτές οι περιοχές δεν έχουν τόσο μεγάλη δυνατότητα διαφοροποίησης, οικονομικής διαφοροποίησης όπως άλλες περιοχές. Δεν έχουν τη δυνατότητα μεγάλων και ταχύτατων αναδιαρθρώσεων όπως σε άλλες περιοχές η διαφοροποίηση είναι πολύ ε, πιο περιορισμένη, οι δυνατότητες, ε, το φάσμα δυνατοτήτων είναι πολύ πιο ε, περιορισμένο και η ανάπτυξη είναι αργή και άρα δεν μπορούμε να αφήσουμε τέτοιο κενό με αυτόν τον αρνητικό αντίκτυπο. Θα εγκαταλείψουν όλοι τα νησιά αυτά. Κατόπιν οι αζόρες. Οι αζόρες παράγουν κυρίως γάλα και κρέας κρέας ε, που πλήττεται τελείως από αυτή τη σύμφωνια με το Μερκοσούρ ε, και το γάλα. Ξέρετε ότι έχει ανακοινωθεί η κατάργηση των γαλακτοκομικών ε, ποσοστώσεων. Άρα θα πρέπει κάπως να αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες προκλήσεις. Ο Γκαμπρίλ Μάτο τις προσδιορίζει επαρκώς, εισηγείται σωστά μέτρα, αλλά η αηφορία των μέτρων θα πρέπει να συνδυαστεί με ενισχυμένο και ευέλικτο προϋπολογισμό. Άρα απευθύνω έκκληση προ όλου, παρακαλώ, να δείξετε ιδιαίτερη ευαισθησία προς αυτές τις ζωτικού χαρακτήρα ανάγκες που έχουν ε, αυτές οι περιοχές και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις από αποκεντρωτέ περιοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Πατράο Νέβε. ο κύριος Μέγε. Ευχαριστώ, Η έκθεση αυτή ε, αναμφισβήτητα είναι εξαιρετική ως προς το περιεχόμενο και συγχαρητήρια γιατί συμπεριλαμβάνει και πάρα πολλά σημαντικά θέματα ουσίας. Αλλά ως νομικός πρέπει να πω ότι και το δευτερεύον γίνεται καμιά φορά πρωτεύον. Γι' αυτό το γερό στις άμεσες ενισχύσεις και στην ανάπτυξη υπαίθρου ο πρόεδρος Παόλο και εγώ ε, ελέγχουμε σε ποιο βαθμό η κατεξουσιοδότηση πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή οι εκτελεστικές ε, πράξεις πρέπει να ε, ανατεθούν. Είναι πολύ σημαντικές οι η πράξη και θα είναι όλο και περισσότερο για το Κοινοβούλιο γιατί μπορούμε να έχουμε λόγο και στην εφαρμογή. Κάτι που μέχρι τώρα ε, μας ε, είχαν ε, αρνηθεί λόγω τη επιτροπολογίας. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό. Στην έκθεση αυτή σε πολλέ τροπολογίε ε, πρόκειται για πολλέ εκτελεστικές πράξεις ή κατεξουσιοδότηση. Και το κοίταξα λίγο είναι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, και όποτε ζητάει εκτελεστικές πράξεις ή κατεξουσιοδότηση ακολουθήσατε αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνατε κάποιες τροποποιήσεις αλλά δεν ζητήσετε να αλλάξουν οι πράξεις ε, παρακαλώ να το δούμε επί της ουσίας αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτελεστικές πράξεις πρέπει να είναι όντως εκτελεστικές ε, γιατί εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την κατάσταση. Θα τα αφήσουμε έτσι ή μήπως θα ζητήσουμε να είναι κάτι εξουσιοδότηση ας πούμε για να είμαστε παρόντες ε, και στην εκτέλεση. Δεν χρειάζεται να το υιοθετούμε αυτούσιο αυτό όπως το προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί της ουσίας να το ξανακοιτάξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μάιερ. Είναι σημαντικό διότι θα πρέπει να διατηρήσουμε μία οριζόντια προσέγγιση και να είμαστε ομοιογενείς σε όλες τις νομικές πράξεις προσαρμογής με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο Σέρχιο Γκουτιέρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό, για να μην είμαι επαναληπτικός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μάτο, τον εισηγητή, για την ε, δουλειά του σε αυτή την έκθεση όπως επίσης και την προσωπική φιλοδοξία, την προσωπική φιλοδοξία που ανέφερε και ο κύριος Άλβες, ο Παύλο Άλβες και τον ευχαριστώ. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα, τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του ΠΟΣΕΙ, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις περιοχές, περιοχές, για τις νησιωτικές περιοχές, για τη ζάχαρη, για την ντομάτα, για τις μπανάνες, αλλά κυρίως για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δήλωση. Δεν μιλάμε εμείς εδώ μόνο για γεωργία ή ειδικέ βοήθειες σε περιοχές που έχουν δυσκολίες, που να παράγουν, να ανταγωνιστούν όπως έλεγε ο εισηγητής αλλά συν δηλαδή και τα προβλήματα, τα φυτοϊγειονομικά προβλήματα, όπως έλεγε ο εισηγητής. Μιλάμε και για τομέα που παίζει σημαντικότατο ρόλο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Εγώ υποστηρίζω απόλυτα ότι, θα, ότι είναι ανεπαρκές το 20% αύξησης της πρικοδότησης στον προϋπολογισμό του ΠΟΣΕΗ. Αν θέλουμε εμείς να είμαστε πιο φιλόδοξοι, θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και όσον αφορά στο δημοσιονομικό δελτίο και στη συγχρηματοδότηση. Και η σοσιαλιστική ομάδα ζητά να βελτιώσουμε τους ελέγχους ε, στα σύνορα τροποποιώντας και το σχετικό κανονισμό εάν χρειάζεται. Αυτά ήθελα να πω. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σιώδη Σιγητή αλλά και τον κύριο Μάτο. Ευχαριστώ κύριε Γκουτιέρες. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο Διευθυντής, ο κύριος Μπότσαρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριος Μποσάχ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι και για μένα και για την Επιτροπή παίζεται η αξιοπιστία της ΚΑΠ. Δηλαδή, παίζεται ακριβώς στο κατά πόσο η ΚΑΠ λαμβάνει υπόψη της τις ειδικές ανάγκες των πιο ευπαθών περιοχών της Ένωσης. Και οι απομακρυσμένες ε, περιοχές της Ένωσης εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία. Γι' αυτό θέλει η Κομισιόν να έχει μια συνεκτική και αποτελεσματική πολιτική για να διασφαλίσει την γεωργική παραγωγή σε αυτές τις περιοχές. Όσον αφορά στις τροπολογίες του κυρίου Μάτο του εισηγητού. Θα ήθελα σύντομα να σας αναφέρω τα πιο σημαντικά σημεία για την νομοθετική βάση άρθρου 349. Δεν θα έχει αντιρρήσεις η Κομισιόν να χρησιμοποιήσουμε αυτή την νομοθετική βάση, διότι μπορούμε να πούμε σαφώς ότι αποτελεί την βάση για την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των απομακρυσμένων περιοχών. Τώρα για το λόγο, για το σήμα δηλαδή των ε, υπερπεριφερειακών περιοχών πάνω στα προϊόντα και εδώ συμφωνώ. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στην, γραμματεία, στην διεύθυνσή μου εγκρίναμε ένα πρόγραμμα ούτως ώστε να δημοσιοποιήσουμε το λόγο αυτό, το σήμα αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα χρηματοδοτήσουμε αυτή την προπαγάνδα με 11 εκατομμύρια ευρώ. Και βλέπετε ότι η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει. Για τις ασφαλίσεις, τις γεωργικές ασφαλίσεις θα πρέπει να περιμένουμε την γενική συζήτηση που θα γίνει για ένα δίκτυ προστασίας των γεωργών και η, η ασφάλιση και η συγχρηματοδότηση της ασφάλισης είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για όλους τους γεωργούς. Και φυσικά για τους ε, γιοργούς ε, των ε, ακραίως απομακρυσμένων περιοχών. Για να καλύψουμε αυτές τις ασφαλίσεις πρέπει να υπάρχουν και κρατικές ενισχύσεις. Αλλά το να, γίνει, να είναι ενίσχυση μόνο κρατική, εμάς μας δημιουργεί νομικά προβλήματα. Τώρα για, τα υπόλοι, για υπόλοιπες τοποθετήσεις, ε, πέρα από αυτά που είπε ο κύριος Μάτο, ακούσαμε να γίνεται λόγος ε, για τις επιπτώσεις των διεθνών συμφωνιών στην παραγωγή. Είναι σαφές ότι θα πρέπει εμείς να περιφρουρήσουμε ούτω ώστε οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες να μην έχουν καταστρεπτικές επιπτώσεις αυτές τις περιφέρειες ε, και στη γεωργική τους παραγωγή. Αλλά όπως είπε ο κύριος Μάτο, ε, το να προχωρήσουμε σε μια αυτόματη αντιστάθμιση, ε, για να καταλήξουμε σε αυτό έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Εμείς ε, η Κομισιόν δεν θέλει μια αυτόματη αποζημίωση, αντιστάθμιση, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως διαπιστώσαμε και στη συμφωνία για τις, για, συμφωνίες για την μπανάνα, το να έχουμε, να αποδείξουμε την απευθείας ε, σχέση μεταξύ, ε, μεταξύ αιτίας και αιτιατού. Είναι δύσκολο λοιπόν εμείς να εισάγουμε ένα τέτοιο μέσο. Τώρα ενδυνάμει η εκτίμηση των επιπτώσεων μιας διεθνούς ε, εμπορικής συμφωνίας ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να το κάνει η Κομισιόν. Επίσης κύριε Μάτο αναφέρατε τις παραδοσιακές ποσότητες. Ζητήσατε να υπάρξει μία ενημέρωση. Και εδώ η Κομισιόν ε, ήταν κάπως εχθρική σε αυτό. Διότι πάντοτε εμείς ανησυχούσαμε να μην ανοίξουμε το, το κουτί της κερδοσκοπίας. Αν συμφωνήσουμε ότι το κάνουμε γιατί εμείς ε, πριν από 20 χρόνια ορίσαμε αυτές τις ε, παραδοσιακά παραγόμενες ποσότητες, ε, σίγουρα τότε μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αλλά εκείνο το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να δεχθεί η Κομισιόν είναι να γίνεται αυτή η ενημέρωση ετησίως ή κάθε δύο χρόνια διότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κερδοσκοπία. Φυσικά 20 χρόνια είναι ιδιαίτερα μακριά περίοδος και μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει, να διορθώσουμε λοιπόν τις ποσότητες. Για τις ε, προκαταβολές. Να σας παραπέμψω στη γενική συζήτηση, γιατί μέσα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ παίζεται όλο το θέμα της, ε, προκαταβο... της ε, καταβολής των πληρωμών, των προκαταβολών, συγγνώμη. Δεν υπάρχει κανένας ε, λόγος αν τελικά συνεχίσουν να ισχύουν οι προκαταβολές να μην τις δίνουμε και στην περίπτωση των απόκεντρων περιοχών. Τώρα για τον προϋπολογισμό δεν είναι δουλειά μου να το συζητήσω εδώ μαζί σας. Εγώ απλώς μπορώ να το σημειώσω, να σημειώσω τις επιθυμίες σας και να προσθέσω κονδύλια στον δημοσιονομικό φάκελο ε, της γεωργίας αυτές τις περιοχές. Τώρα, αν τα κονδύλια Αν πρέπει λοιπόν να δοθούν κονδύλια, θα πρέπει αυτά τα λεφτά να τα βρούμε από αλλού από άλλους τομείς, από άλλους ε, γεωργούς. Είτε θα πρέπει αυτό το χρήμα να έρχεται απ' έξω. και όχι από το γεωργικό προϋπολογισμό. Αυτά πρέπει όμως να τα δούμε σε πολιτικό και δημοσιονομικό επίπεδο. Κυρία Γκαρσία, ρωτήσατε αν μου παρουσίασαν τη μελέτη, ναι. Είναι η απάντησή μου. Την προηγούμενη εβδομάδα δύο ώρες πάνω κάτω έφαγα για την παρουσίαση της ε, μελέτης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικοδομητική μελέτη. Είναι μια μελέτη η οποία... εξετάζει το θέμα του κόστους. Ξέρουμε ότι το κόστος είναι ψηλότερο σε αυτές τις περιοχές. Και εξετάζει επίσης και τη σχέση εισοδήματος και κόστους. Και πραγματικά βρισκόμαστε στο χείλο του γκρεμού από ό,τι φαίνεται. Αλλά διότι διαπιστώνουμε ότι είναι ελάχιστο, ελάχιστο το περιθώριο κέρδους του Γιώργου. Και η μελέτη αυτή δεν στέκεται μόνο στον τομέα της μπανάνας, αλλά λαμβάνει υπόψη τη γεωργική παραγωγή στις απομακρυσμένες περιοχές. Και θα μας βοηθήσει να αποφασίσουμε πόσο χρήμα θα πρέπει να βάλουμε στον δημοσιονομικό φάκελο για να διασφαλίσουμε τη γεωργική δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές. Αλλά ξέρετε όμως εγώ σε αυτό το στάδιο δεν μπορώ εγώ να κρίνω κάτι γιατί δεν είναι στα δικά μου επίπεδα αυτές οι αποφάσεις. Κύριε Αλβές, εσείς ε, μιλήσατε για το 20% για το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού. Εμείς ως Κομισιόν Εμείς όμως θέλουμε να είμαστε σε μια δημοσιονομική ουδετερότητα. Θέλουμε να δώσουμε ευελιξία στα κράτη-μέλη αλλά η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει μια δημοσιονομική ουδετερότητα, ενώ οι συνάδελφοί σας και εσείς θα θέλατε να υπάρξει μια προσάυξηση του ποσού στον γενικό προϋπολογισμό. Αλλά αυτό πάλι σας είπα είναι μια απόφαση που δεν είναι στα δικά μου επίπεδα και δεν μπορώ να πω τίποτε εγώ. Κύριε Μάγερ, τονίσατε την σημασία της ε, κατά περίπτωση κρίσης των εξουσιοδοτημένων πράξεων ή των εκτελεστικών πράξεων. Εγώ νομίζω ότι έχετε δίκιο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνετε. Εγώ ως Κομισιόν μπορώ να πω ότι στον κανονισμό Ποσέη έχουμε ακολουθήσει τη γενική προσέγγιση της Κομισιόν που θα την βρείτε και στους ε, μεγάλους ε, κανονισμούς ε, της, των, της κοινής οργάνωσης των αγορών. Πάντοτε εκεί κρατήσαμε την ίδια προσέγγιση, την ίδια στάση και την εφαρμόσαμε και στον κανονισμό Ποσέη. Και δεν το κρύβω, η προσέγγιση της Κομισιόν εντάσσεται μέσα στη γενική έμπνευση προστασίας των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου και στοχεύει στην πιο στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Βέβαια πρέπει να προχωρήσουμε σε μία κατά περίπτωση εξέταση για να δείτε αν σας βολεύει και η πρόταση της Κομισιόν. Ε, ευχαριστώ κύριε Διευθυντά, ευχαριστώ την Κομισιόν. Τον τελικό λόγο έχει ο κύριος Μάτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πάρα πολύ σύντομα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την τοποθέτησή τους και την Κομισιόν και να ολοκληρώσω λέγοντας πράγματι Πρόκειται για μια φιλόδοξη έκθεση αλλά είναι απόλυτα ρεαλιστική και το κάθε μέτρο το οποίο προτείνουμε είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Έλαβε υπόψη αυτή η έκθεση τις γνώμες όλων και φυσικά είναι και ανοιχτή και στις ε, άλλες τροπολογίες που θα έρθουν. Βέβαια πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το θέμα των εκτελεστικών πράξεων και των εξουσιοδοτημένων πράξεων. Των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Εγώ ευχαριστώ και τον ε, Διευθυντή διότι φαίνεται ότι τελικά ακολουθούμε ίδιους δρόμους. Έχουμε περισσότερα σημεία που μας ενώνουν από τη σημεία που μας χωρίζουν. Είμαι πεπισμένος ότι και ο Διευθυντής αλλά και η Κομισιόν συνολικά πιστεύουν ότι οι ακραίως απομακρυσμένες περιοχές αποτελούν μια ευκαιρία για την Ευρώπη. Και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι τα λίγα προβλήματα τα οποία εκκρεμούν, ακόμη και στο θέμα δηλαδή της χρηματοδότησης, θα μπορέσουν να αιτιολογηθούν σωστά και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γκαμπριέλ. Θυμίζω σε όλους τους συναδέλφους ότι 11 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και 19 Σεπτεμβρίου θα ψηφιστεί η έκθεση. Πάμε στο σημείο 5 στην ημερήσια διάταξη. Ειδικά μέτρα στον τομέα της Γεωργίας υπέρ των μικρών νησιών του Αιγαίου. Ο Γιώργος Παπαστάμκος είναι ο εισηγητής. Η συζήτηση για το σχέδιο έκθεσης ε, του κυρίου Παπαστάμκου αφορά στον, στην πρόταση κανονισμού, στον κανονισμό της γνώμη της Κομισιόν για τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Πρόκειται για τον 1405-2006 του ε, Συμβουλίου ε, ειδικά μέτρα για τη Γεωργία, για τα μικρά νησιά. Αυτός ο κανονισμός έχει τροποθεί πολλές φορές και η Επιτροπή ζήτα να διορθωθεί. Και είναι παράλληλη αυτή η πρόταση και με την ε, συζήτηση που είχαμε προηγουμένως ε, για τις ε, απομακρυσμένες περιοχές. Τα μικρά νησιά του Αιγαίου αποτελούν τεράστια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εδαφική συνοχή. Δίνω το λόγο ευθύ αμέσως στον κύριο Παπαστάμκο και Γιώργο έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα κύρια σημεία της αιτιολογικής έκθεσης επί της συγκεκριμένης προτάσεως κανονισμού τη Κομισιόν τα παρουσίασα σε προηγούμενη συνεδρία τη Επιτροπή μα. Παραλείπω να αναφερθώ εκ νέου στα σημεία αυτά. Έτσι θα είναι πάρα πολύ συνοπτικέ οι παρεμβάσει μου, οι παρατηρήσει μου επί της πρόταση κανονισμού τη Επιτροπή σχετικά με το καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Και αυτέ οι σύντομε παρατηρήσει μου εκκινούν από δύο επισημάνσεις. Καταρχάς εξετάζουμε σήμερα την ομοθετική πρόταση που έχει χαρακτήρα αναδιατύπωσης, recast και όχι αναθεώρησης. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, θα πρέπει να αναμένουμε προς τα τέλη του 2011 έκθεση αποτίμησης, αξιολόγησης της εφαρμογής του καθεστώτος, στην οποία θα βασιστεί νέα νομοθετική πρωτοβουλία με ουσιαστικού περιεχομένου μεταβολές. Η δεύτερη επισήμανση, σύμφωνα με το δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει την πρόταση κανονισμού, οι πόροι του καθεστώτος εγγράφονται σε δύο γραμμές του κοινοτικού προπολογισμού που ανήκουν στον πρώτο πυλώνα, δηλαδή τι άμεσε ενισχύσει τη κοινή αγροτική πολιτική, συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγύσεων ως άνω ε, δύο ε, παρατηρήσεις αρχής οριοθετούν το πλαίσιο των προτάσεών μου που μπορούν να συνοπιστούν στα ακόλουθα ε, έξι σημεία. Πρώτο σημείο, αύξηση κατά 30% των κονδυλίων που προορίζονται για το καθεστώς των μικρών νησιών του Αιγαίου. Δεύτερο σημείο, δυνατότητα μεταφοράς των αδιαθέτων ποσών μεταξύ των ειδικοτέρων μέτρων που προβλέπονται στο καθεστώς καθώς και δυνατότητα μεταφοράς των ετησίως αδιαθέτων ποσό στο επόμενο έτος. Τρίτο σημείο, σε ό,τι αφορά το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού, ε, ε, ε, να υπάρχει επέκταση της επιδότησης πέραν του εφοδιασμού σε πρώτες ύλε και στην μεταφορά των παραγωμένων αγροτικών προϊόντων πρωτογενών ή μεταποιημένων από τα νησιά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέταρτο σημείο, περισσότερο ενεργή συμμετοχή και συμβολή των αρμοδίων περιφερειών και δήμων, ε, δηλαδή της τοπικής κοινωνίας, τον, ε, στον καταρτισμό των προγραμμάτων εφαρμογής του καθεστώτος. Πέμπτο σημείο, να υπάρχει σύνδεση της καταβολής ενισχύσεων με την παραγωγή σε μια μελλοντική ουσιαστικού περιεχομένου αναθεώρηση του καθεστώτος. Και έκτο και τελευταίο σημείο, ε, προβλέπεται, προνοείται προτείνω την ομοιόμορφη διατύπωση των λεγόμενων τυποποιημένων διατάξεων κατ' εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ των, των θεσμικών οργάνων κατ' εφαρμογή της διαθεσμικής ή διοργανικής συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Παπαστάμκο. Ο Αντιπρόεδρος Πόλσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Περιμένω λίγο για να βάλουν όλοι τα ακουστικά. Ε, Προτιμώ να μιλάω ειδικά. Είναι πάρα πολύ καλή η έκθεση που εξετάζουμε και χαίρομαι που την ανέλαβε ο Παπαστάμκος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα ανεξάρτητα από το θέμα των εξόχως απόγκεντρων περιοχών. Όλες αυτές οι μειονεκτικές περιοχές, οι περιοχές που μειονεκτούν σε σχέση με τις υπόλοιπες, έχουν κάτι κοινό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι αυτό, οι συνθήκες είναι τέτοιες ώστε είναι πάρα πολύ δύσκολο να οικοδομήσουμε μία εξορθολογισμένη γεωργία μεγάλης κλίμακος. Και δεν συζητούμε μόνο για τον συνολικό ανεφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωτίστως αυτό που επιθυμούμε είναι να διατηρήσουμε τον πολιτισμό και την ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, για την χρήση και καλλιέργεια της γης. Ε, ε, Ε, είτε μιλάμε για την καλλιέργεια στα νησιά του Αιγαίου με τις αναβαθμίδες, ε, είτε μιλάμε για άλλες ε, μορφές καλλιέργειας που χρησιμοποιούνται στη μέση του ωκεανού. Ανεξαρτήτως περιοχής πρέπει να προστατεύσουμε αυτές τις περιφέρειες γιατί φέρουν πολιτισμό. Είτε μιλάμε, ξαναλέω, για το περιβάλλον, είτε για τις καλλιεργητικές μεθόδους, είτε για τα ίδια τα τρόφιμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και χρειάζεται υποστήριξη από όλους, ώστε αυτές οι περιοχές ε, να προστατεύσουν ε, τα μικρότερα επαγγέλματα γιατί είναι μηχανοργανωμένοι σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό η παραδοσιακή βιομηχανία είναι όλα εξορθολογισμένα, γίνεται σωστά ανεφοδιασμός, η παραγωγή κτλ. Ναι, σωστά όλα αυτά, αλλά χρειαζόμαστε τις βασικές γνώσεις που είναι η προϋπόθεση, οι βασικές παραδοσιακές γνώσεις που είναι η προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ε, βιομηχανίας. Ε, και λόγω της ζωτικής σημασίας που έχουν αυτές οι γνώσεις για τις ε, μειονεκτούσες ε, περιοχές. Κάτι άλλο που επίσης ε, συνιστά κοινό σημείο για όλες αυτές τις εξόχως τις περιοχές ε, είναι το θέμα των μεταφορών και της διασύνδεσης. Ε. Το θέμα της λογιστικής μελητία Είναι θέμα επιβίωσης για τους κατοίκους αυτών των περιοχών και εδώ δεν έχει καμία σημασία το τοπικό χαρακτηριστικό. Ποιο είναι το τοπίο, ποια είναι τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, ποια είναι τα παραδοσιακά τρόφιμα. Μα δεν έχει καμία σημασία. Είτε μιλάμε για τον ε, απομακρυσμένο βορρά, για τις δαστώσεις περιοχές, είτε μιλάμε για τις νησιώτικες περιοχές του Αιγαίου. Αυτό είναι ένα κοινό σημείο. Οι μεταφορές και οι παραδόσεις. Αυτά είναι τα δύο βασικά σημεία. Ευχαριστώ Αντιπρόεδρε Πόλσον. Ο κύριος Δανέλης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο οι παρατηρήσεις και οι διαπιστώσεις της ε, Αντιπροέδρου και ε, συμφωνώ απολύτως ότι είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για το ευρωπαϊκό επικοδόμημα η αντιμετώπιση των νησιωτικών περιφερειών της ε, Υπήρου μας. Και βεβαίως το θέμα αυτό έχει ευθεία σχέση με αυτό που συζητήσαμε αμέσως πριν. Ε, να πω επίσης ότι δεν είναι κοινό τόπος, δεν είναι ε, κοινά αποδεχτό ότι οι συνθήκες διαβίωσης αλλά και κυρίως οι συνθήκες ανάπτυξης των νησιών διαφέρουν πάρα πολύ από τις υπηρετικές περιοχές. Αυτό δεν είναι αυτονόητο, παρά μονάχα αν διαθέτεις κάποια βιωματική σχέση με νησιά. Δεν είναι μονάχα οι πολύ δύσκολες δημογραφικές πιέσεις δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικά ε, μοντέλα ανάπτυξης πέρα από τις οριακής σε πολλές περιοχές γεωργίας ή κτηνοτροφίας και του τουρισμού, που πολλές φορές όμως έρχονται και σε αντιπαράθεση αυτή, οι, αυτές οι αναπτυξιακές προσπάθειες εξαιτίας του ανεπαρκούς νερού, ας πούμε, ή της διαχείρισης του εδάφους. Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα της δυσκολίας πρόσβασης και τα κόστη είναι πολύ σημαντικότερα όπως επίσης τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς για απροσδιόριστο χρόνο μπροστά μας έχουμε τις αυξημένες πιέσεις της λαθρομετανάστευσης. Ε, για όλους αυτούς τους λόγους ε, αξίζει τον κόπο να ε, σκύψουμε πάνω στις ανάγκες ανάπτυξης των νησιών με ένα διαφορετικό τρόπο. Ε, όσον αφορά την γεωργία ή την κτηνοτροφία, το να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη βιοπικιλότητα, να μπορέσουμε να στηρίξουμε το τοπικό γενετικό υλικό, ε, το οποίο είναι και βεβαίως πολύ πιο ε, προσαρμοστικό στις ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες της κλιματικές ή την ε, λειψιδρία ή την, τους έντονους ανέμους και ούτω καθεξής είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση και ένα χρέος. Ε, όπως είπε ο συνάδελφος ο Παπαστάμκος με τον οποίο έχουμε μια στενή συνεργασία ε, και τον ευχαριστώ για αυτό η, δεν συζητάμε τώρα για την αναθεώρηση του κανονισμού ίσως έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε στο τέλος του χρόνου όμως με την ευκαιρία αυτής της προσαρμογής στην ε, Λισαβόνα νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σημειώσουμε την αναγκαιότητα της αύξησης του ε, ποσού χρηματοδότησης αυτού του κανονισμού, πράγμα το οποίο επισημαίνεται εξάλλου και από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, ε, και επίσης να απαλείψουμε αυτό που έναν κανονισμό που δεν καταλαβαίνω, δεν νομίζω ότι έχει σχέση με λογική, το να μην ε, χρηματοδοτούνται, να μην ε, ε, στηρίζονται και οι μεταφορές των γεωργικών προϊόντων από τα νησιά προς την υπηρετική χώρα. Δεδομένης της μοναδικότητας και της ποιότητας των προϊόντων αυτών και με δεδομένο το ότι δεν υπάρχουν ανεπτυγμένα δίχτυα εσωτερικής αγοράς και πρόθεση των προϊόντων και κατανάλωσής τους επιτόπου, νομίζω ότι θα πρέπει να απαλληφθεί αυτή η διάταξη από το σημερινό κανονισμό. Ε, ευχαριστώ πολύ και θα επανέλθουμε στην συνέχεια της κουβέντας μας ε, όταν τα πράγματα είναι και πιο όριμα. Ευχαριστώ. Κύριε Δανέλη, Τζοβάνι Λαβία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Παπαστάμκο για την εξαιρετική εργασία του μας ε, δίνει νέες προπτικές και διαφωτίζει με νέο τρόπο όλο αυτό το καθεστώς ενισχύσεων για τα νησιά του Αιγαίου. Σημερίζουμε πλήρως τα έξι σημεία τα οποία υποβάλλει στην προσοχή μας στο τέλος της έκθεσής του. Θα ήθελα όμως, αν μου επιτρέπετε, να τονίσω δύο ε, ε, πλευρές και να ρωτήσω δύο πράγματα. Από τη μια ο συνάδελφος Παπαστάμκος ζητά αναθεώρηση του δημοσιονομικού καθεστώτος. Αυτό προβλέπει βέβαια και εμπλοκή των αρχών του προϋπολογισμού που δεν προβλέπεται εδώ στην... Ε, δεν υπάρχει τίποτα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για αυτή την έκθεση. Το δεύτερο αφορά στην Επιτροπή και η οποία είναι και επακόλουθη της ερώτησης που είχα παρουσιάσει στην προηγούμενη Ολομέλεια και που αφορά στα νησιά της Σικελίας τα οποία χαρακτηρίζονται από την ίδιες συνθήκες περιφερικότητας και νησιωτικότητας. Πρόκειται για νησιά τα οποία δέχονται μεταναστευτικά φαινόμενα, των οποίων η γεωργία έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την υπερπεριφερειακότητα, όπου το κόστος παραγωγής είναι σαφώς υψηλότερο από ό,τι στην υπηρετική χώρα και όπου και το κόστος των προϊόντων είναι πολύ υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη παραγωγική πραγματικότητα στην Ευρώπη. Την προηγούμενη φορά στην Επιτροπή Γεωργίας η Κομισιόν μας είχε πει ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στον να εφαρμοστεί ένα αντίστοιχο καθεστώς και για αυτά τα νησιά. Φτάνει να υποβληθεί έτοιμα από το κράτος μέλος. Τώρα ενημερώνω την Κομισιόν ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει υποβάλει τη σχετική αίτηση σήμερα πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε για την διαμόρφωση αυτού του νέου καθεστώτος. Θα πρέπει να επεκτείνουμε τον, το καθεστώς των μικρών νησιών του Αιγαίου ή πρέπει να φανταστούμε ένα νέο καθεστώς. Ευχαριστώ κύριε Λαβιέ. Αν δεν υπάρχει το λόγο, ο Διευθυντής ε, έχει το λόγο και μετά ο κύριος Παπαστάμκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι ακόμη πιο σύντομος αυτή τη φορά. Ό,τι ανέφερα σχετικά με το ΠΟΣΕΙ, μουτά της μουτάντης εφαρμόζεται και σε αυτή την έκθεση. Ο κύριος Παπαστάμκος έχει δίκιο καταρχήν. Πρόκειται για μία αναδιατύπωση και δεν θα πρέπει να ε, περιμένετε πολύ. Και εμείς εδώ ολοκληρώνουμε την ε, έκθεσή μας και όπως είπε και ο κύριος Παπαστάμκος θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει τα διάφορα σημεία λεπτομερώς. Εδώ και πάλι όσον αφορά στην αύξηση κατά 30% όπως το είπα και προηγουμένως, συμφωνούμε καταρχήν, αλλά και αυτό πάντα στα πλαίσια της δημοσιονομικής ουδετερότητας. Τώρα κύριε Παπαστάμκο για την ιδέα σας για να, μετα, μεταφερθούν τα μη ε, χρησιμοποιημένα κονδύλια από το χρόνο νη στον χρόνο νη συνένα, εκεί θα έχουμε πρόβλημα, διότι έχουμε ετήσιους προϋπολογισμούς. Και αυτό θα δημιουργήσει ένα κάποιο πρόβλημα στην ευθυγράμμιση της ιδέας με τους δημοσιονομικούς κανόνες όπως υπάρχουν, όπως ισχύουν σήμερα, που είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Κυρία Πόλσεν, προσυπογράφω την κάθε σας λέξη και τον τρόπο με τον οποίο τονίσατε τη σημασία αυτών των νησιών και των υπερπεριφερειακών περιοχών και μάλιστα εκτίμησα ιδιαίτερα ότι δεν περιοριστήκατε μόνο στην ε, γεωργική παραγωγή, όπως έκανα και εγώ εξάλλου προηγουμένως, μιλήσατε για, την για τον σύνδεσμο μεταξύ παραγωγής και κουλτούρας ε, στο νησί. Αποτελεί η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρήκατε τα λόγια που χρειαζόντουσαν για να περιγράψετε το μέγεθος της πρόκλησης για την εξέβρεση της σωστής πολιτικής ούτως ώστε να μπορέσουν να μακροβιώσουν όλες αυτές οι περιφέρειες. Αναφέρατε και τις μεταφορές. Μα φυσικά, αν λάβουμε υπόψη και τη γεωγραφική κατάσταση αυτών των περιοχών, φυσικά είναι ένα πρόβλημα αλλά η μεταφορά από την υπηρετική χώρα στα νησιά ρυθμίζεται. Χρησιμοποιούμε τα κονδύλια του ΕΡΕΣΑ. Εκεί όπου όμως ε, υπάρχει ακόμα δυνατότητα είναι οι τοπικές μεταφορές, οι μεταφορές μέσα στο νησί όπου δεν είναι τα ΕΡΕΣΑ που παίζουν, αλλά η υποστήριξη στην τοπική παραγωγή και θα πρέπει εμείς να προσαρμόσουμε τη διατύπωση ενός ε, τίτλου στο, του καθεστώτος για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και αυτόν τον τομέα. Κύριε Δανέλη, και εσείς περιγράψατε πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο μας ε, χρειάζεται για να ολοκληρώσουμε τον κοινό μας στόχο. Το από το 2000 ε, ό,τι έχουμε ε, μέχρι σήμερα κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να διατηρήσουμε την ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής και της κάθε παραγωγής ε, δημιουργώντας και το σχετικό δημοσιονομικό φάκελο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε παραπάνω και να βρούμε τα απαραίτητα μέσα για να καταπολεμήσουμε επιτόπου τα προβλήματα, όπως και εσείς ο ίδιος αναφέρατε. Αυτό έχει να κάνει και ε, κυρίως με την ετήσια μας έκθεση παρά με την τωρινή αναδιατύπωση. Και κύριε Λαβία τώρα, ναι, θυμούμε πάρα πολύ καλά όταν είχα αναφέρει ότι η Ιταλία θα έπρεπε να προχωρήσει σε αυτό το διάβημα εμένα όμως δεν μου ήρθε ακόμη αυτή η αίτηση στο γραφείο μου. Δεν μπορώ να σας πω σήμερα αν το καλύτερο μέσο είναι ένα ειδικό καθεστώς ή αν θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε αυτό το καθεστώς με τα νησιά του Αιγαίου. Θα μπορούσαμε, ναι, το λέω έτσι αυθόρμητα τώρα στη στιγμή. Τώρα, εάν τα προβλήματα τα οποία ισχύουν για τα νησιά γύρω από τη Σικελία είναι παράλληλα με εκείνα των μικρών νησιών του Αιγαίου, τότε γιατί όχι. Να διευρύνουμε το, εφαρμοσ... το γεωγραφικό εφαρμοστικό πεδίο. Αυτό όμως απαιτεί εις βάθος εξέταση και πώς ε, θα, το... θα προχωρήσουμε. Θα γίνει πρώτα μία εσωτερική εξέταση και μετά αν έχουμε προβλήματα ή συμπληρωματικές ερωτήσεις ε, θα διαβουλευτούμε με τις Ιταλικές αρχές. Και στο τέλος ε, θα υποβάλουμε μία πρόταση για να διευρύνουμε ένα υπάρχον καθεστώς ε, και να καταλήξουμε μετά σε προτάσεις ή με ειδικό καθεστώς για τα προβλήματα των νησιών γύρω από τη Σικίλια. Γιατί φυσικά και για αυτά τα νησιά θα πρέπει να εγγυθούμε την επιβίωσή τους. Ευχαριστώ κύριε Διευθύντα. Ο κύριος Παπαστάμκος για να ολοκληρώνει. Γιώργο έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Αντιπρόεδρο, την κυρία Πόλσεν για τις παρατηρήσεις της. Πάρα πολύ ε, ε, δημιουργικές παρατηρήσεις της και αυτή την ξεχωριστή ανάγνωση που κάνει ε, σε ό,τι αφορά την κατάσταση της γεωργίας στα μικρά νησιά του Ηλιό και σε νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης, όπως επίσης και τον κύριο Δανέλη και τον κύριο Λαβία για τις ε, πολύ γόνιμες ε, συνεισφορές τους και καθώς και τον εκπρόσωπο, όλος ιδιαίτερος τον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν. Και στέκομαι λίγο σε αυτό που είπε η κυρία Πόλσεν, η κυρία Αντιπρόεδρος, και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η έννοια της γεωργικής δραστηριότητας κατά την πλέον σύγχρονη σύλληψή της σε νησιωτικές περιοχές όπως αυτή των μικρών νησιών του Αιγαίου ε, συγκοινωνεί αναπόδραστα με την αηφόρο οικονομική, κοινωνική και οικολογική ανάπτυξη. Και κωδικοποιώ αυτό που είπε η κυρία Πόλσεν με τη διατήρηση συνεπώς του φυσικού και πολιτισμικού τοπικού πλούτου, της παράδοσης, του πολιτισμού. Και μια παρατήρηση ακόμα σε ό,τι αφορά τα νησιά του Αιγαίου. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η διασπορά των νησιών και η ομαδοποίησή του σε αρχιπέλαγος αποτελούν εμπόδια για τον εφοδιασμό και το εμπόριο, αυξάνοντας κατακόρυφα τα έξοδα ε, μεταφοράς. Τα εφιστάμενα δίκτυα μεταφορών χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια και δομικές αδυναμίες και δημιουργώντα ηθίκες διπλής νησιωτικότητας, εφόσον ο εφοδιασμός των μικροτέρων νησιών πραγματοποιείται μέσω άλλων περισσότερο κεντρικών ε, νησιών. Και το περιορισμένο μέγεθος, το εξωτερικός και εσωτερικός δυσπρόσιτον, ο φθήνων και γερασμένος πληθυσμός και έλλειψη βασικών πρώτων υλών, αλλά και δημοσίων αγαθών, όπως είναι το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, όπως και οι γεωφυσικές και κλιματικές συνθήκες, βραχώδες έδαφος, κατακαιρματισμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και ξηρότητα και ισχυρή άνοιμη αντιστοίχω συνθέτουν το εξαιρετικό ιδιόμορφο περιβάλλον των νησιών του Αιγαίου Πελάγος. Και τελειώνω λέγοντας ότι, ε, και χρειάζεται να το υπογραμμίσουμε αυτό, τα νησιά του Αιγαίου αποτελούν εξωτερικό σύνορο της Ένωσης, πέραν δε των ιδιαίτερων δυσχεριών, ε, οι οποίες χαρακτηρίζουν τη γεωργική παραγωγή των μικρών νησιών του Αιγαίου, αποτελούν και δέκτες εξωτερικών μεταναστευτικών, λάθρο μεταναστευτικών πιέσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, τους συναδέλφους για τις συνεισφορές τους και μέσω τροπολογιών όπως θα έρθουν, όπως επίσης και την Κομισιόν για την πάρα πολύ καλή συνεργασία μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Γιώργο. Σας θυμίζω και στην προκειμένη περίπτωση ότι Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 11 Ιουλίου και έγκριση της νομοδότησης 19 Σεπτεμβρίου. Ωραία. Σε αυτό το σημείο πάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Πρέπει να ψηφίσουμε όλοι την κάρτα σας. Αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη. Η κυρία Σάρμπου είναι η συγγήτρια, η Ναπούσα και την αντικαθιστά κύριος Έντσου. Μιλάμε εδώ για τις αγορές των γεωργικών commodities, πρώτων υλών δηλαδή, και η κυρία Σάρβου θέτει προτεραιότητες και τονίζει σημεία που αφορούν στην αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικό τομέα στα πλαίσια της τροφιμικής ασφάλειας. Έχουμε 46 τροπολογίες στη γνωμοδότηση αυτή, όπως επίσης και συμβαστικές τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε λοιπόν εμεί σήμερα στις συμβιβαστικές τροπολογίες και ευχόμεθα η Επιτροπή Ήτρε ως συναρμόδια επιτροπή να προσέξει ιδιαίτερα στη γνωμοδότησή μας. Αν είστε έτοιμοι και αν έχετε όλοι, αν δεν έχετε τη λίστα, να την ετοιμάσουμε. We start with amendment We start with one, amendment 1, two, compromise 1, and if adopted 10, if, if adopted, and etc. Oh, etc. Pronti? Έτοιμοι. Βλέπεις ε, Νίκο, τελικά δεν διαφέρει και πολύ από το μοτετσιτόριο εδώ η κατάσταση. Δηλαδή από το τελικό κοινοβούλιο. Ωραία. Αρχίζουμε. Τροπολογία να μαγκίνες. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψυχοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψυχοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σμιτ. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Εγώ εδώ είμαι και έχω και την κάρτα μου, αλλά δεν δουλεύει. Με πρόδωσε η τεχνολογία. Εντάξει, θα το ελέγξουμε, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Προχωράμε. Τροπολογία 10. Λάιον. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 Νικουλέσκου. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 12. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμό 2. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 18. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 20. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. 20. Απορρίπτεται. 21. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 23 αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. απορρίπτεται. 29. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 30. Ψηφίζουμε. Αρχίζουν οι ψηφοφορίες. Πέρας ψηφοφορίες για την 30. Ψηφίζουμε την 31, αρχίζουν αρχίζει η ψηφοφορία, Πέρας ψηφοφορίας για την 31 εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 4. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5. Αρχής ψηφοφορία, της πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 40. Προσοχή, μιλάμε για τις 40 αρχές ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 41 ψηφίζουμε. 41 πέρας ψηφοφορίας για τις 41 εγκρίνεται. 43 Αρχίζει ψηφοφορία για τη 43, ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 44, Ντάντσιλα, αρχίζει ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 46, Γέγγελ, πέρας ψηφοφορίας για τη 46, εγκρίνεται. Υπήρξε ένα, μια στιγμή suspense, Elizabeth. Και τώρα έχουμε την τελική ψηφοφορία. Αρχίζουμε την ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Σάρμπου. Θα παρακαλέσουμε την κυρία Ίντσου να αναφέρει. Τώρα. Το πιο σημαντικό σημείο στην ημερήσια διάταξη είστε όλοι έτοιμοι. Ο Τζέμς εδώ είναι. Ναι. Τζίμ είσαι έτοιμος. Ωραία. Σημείο 7. Τροποποίηση του κανονισμού 1234 κάθετος 7 του Συμβουλίου όσον αφορά στις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ο εισηγητής είναι ο James Νίκολσον, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πρέπει να ψηφίσουμε τώρα την έκθεση Νίκολσον που αφορά στις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος. Πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, πρόκειται για ένα θέμα συναπόφασης, ένα νομοθετικό σχέδιο. Κατατέθηκαν πάνω από 300 τροπολογίες, αλλά πρέπει να ευχαριστήσω την εξαιρετική δουλειά του εισηγητή μας και όλων των σχεδόν εισηγητών όλων των πολιτικών ομάδων καταφέραμε να βρούμε μια μεγάλη σύγκληση γύρω από 8 συμβιβαστικές τροπολογίες και 19 συμβιβαστικές τροπολογίες τα εκτιμώντας. Λοιπόν, με αυτή την ψηφοφορία εμείς θα δώσουμε εντολή στον εισηγητή να διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο και αυτό εν ώψη της απόλυξης συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση. Πρέπει σήμερα κατά συνέπεια να διαφανεί σαφώς η θέση και οι εμπνεύσεις της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Τζιμ, θες να πεις κάτι? Ναι, θέλω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα καλά σας λόγια. Ελπίζω όταν θα έχουμε τελειώσει ψηφοφορία να είμαστε στην ίδια θέση. Θα ήθελα να τονίσω και πρέπει να πω ότι ήταν ε, δύσκολη υπόθεση και καταλήξαμε ε, σε λίγο σχετικά μικρό αριθμό συμβαστικών τροπολογιών, πράγμα που μας εξέπληξε. Θα πρέπει στην Επιτροπή μας να έχουμε μια συνεκτική θέση για να προχωρήσουμε. Και επευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όλους τους για την πάρα πολύ σκληρή δουλειά τους και πρέπει να σας πω ότι δόθηκαν και σκληρές μάχες ε, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για τους συμβασμούς, αλλά ακόμα και όταν ήταν σκληρά τα πράγματα. Ε, χάρηκα που ήρθατε και εσείς και προεδρεύσατε σε κάποιες από τις συνεδριάσεις και προχωρήσαμε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Πάτρικ και όλο το προσωπικό και τη γραμματεία της Επιτροπής μας ε, που βοήθησαν, αλλά και όλους τους υπαλλήλους των πολιτικών ομάδων που ώρες ολόκληρε αφιέρωσαν, ακόμα και όταν έφευγαν οι βουλευτέ, οι σύμβουλοι έπρεπε να παραμένουν και να συνεννοούνται στο δικό του επίπεδο. Ευχαριστώ λοιπόν όλο το προσωπικό που εργάστηκε στην υπόθεση αυτή και πραγματικά ε, σα συνιστώ να υπερψηφίσετε αυτό το συνολικό πακέτο με τι συμβαστικέ τροπολογίε που επιτύχαμε. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, ευχαριστώ James. Αν είστε έτοιμοι με κάρτα και κατάλογο ψηφοφορίας ξεκινάμε. Να ξέρετε ότι εδώ θα κρατήσει παραπάνω ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τροπολογία 126. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 8. Ψηφίζουμε τον συμβιβασμό 8. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στο συμβιβασμό 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. 171. Στο βάθος της σελίδας 3. Νταντέ. Αρχίζει η ψηφοφορία. 171. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 173. Άλβες. 173. Πέρας ψηφοφορίας. Συμβιβασμός 2. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 205. Ψηφίζουμε την 205. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται θα έλεγα. 210. 210 ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 228 στην επόμενη σελίδα. Αρχίζει η ψηφοφορία. 228 λέει ο πρόεδρος. 228 επαναλαμβάνει ο πρόεδρος. Πέρας ψηφοφορίας. Λοιπόν, Μάρκ, παρακολουθείς ή όχι, γιατί εγώ σας αντιγράφω. Πάμε στον συμβιβασμό 3. Αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία του συγγητή, αριθμός 21. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22. Πάντα του εισηγητή. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται επίσης. Συμβιβασμός 4. Ψηφίζουμε. Ωραία. 238 2-3-8. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. περασε Απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 5. Πώς? Slowly. Μάλιστα. Ε, εντάξει. Τι θέλετε να πείτε. Κυρίσω την ψηφοφορία της τροπολογίας 5. Αυτό είναι το slowly για σας. Ωραία. Ψηφίσατε εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στη σελίδα 10, στην τροπολογία 30. Πρόκειται για τροπολογία του εισηγητή. Ψηφίζουμε για την 30. Ψηφίσατε όλοι, τροπολογία 30. Πέρας ψηφοφορίας. 31. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 39. 39. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβασμός Α. Αρχίζει η ψηφοφορία για τον συμβιβασμό Α. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός Β. Να ψηφίσουμε πρώτα τον συμβιβασμό Β και μετά. Ναι, πρώτα ψηφίσουμε. Ωραία, αρχίζει η ψηφοφορία για τον συμβιβασμό Β. Ψηφίσατε όλοι τον συμβιβασμό Β. Ναι, ε, εγκρίνεται. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σιλβέστρης για μια προφορική τροπολογία. Κύριε Πρόεδρε, έχει μοιραστεί η τροπολογία. Δεν θέλουμε εμείς να επεκτείνουμε τα μέτρα του γαλακτοκομικού τομέα, αλλά θέλουμε απλώς να τονίσουμε ότι υπάρχει και μια τεράστια δυσκολία στην αγορά ελαιολάδου και επιτραπεζίων ελαιών. Η κατάσταση τα τελευταία χρόνια έχει χειροτερέψει πάρα πολύ και σε ορισμένες περιοχές δεν έχουμε ο Γιωργός δεν καλύπτει καν τις δαπάνες ε, παραγωγής. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες και κοινωνικές εντάσεις στον τομέα αυτών. Θα παρακαλούσα λοιπόν η Κομισιόν να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις στα πλαίσια των τριετών προγραμμάτων του 1234 κανονισμού, όπως προβλέπει δηλαδή ο 1234, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα παραμένω σταθερός και λέω ότι δεν θέλουμε να επεκτείνουμε εμείς ε, τα, μέτρα του γαλακτοκομικού τομέα, απλώς ζητάω από την Κομισιόν επί τη ευκαιρία να αναλάβει αυτές ε, τις ε, πρωτοβουλίες. Και παρακαλώ δηλαδή και τον εισηγητή να δεχτεί την προφορική τροπολογία. Εμείς ως Επιτροπή Ασχοληθήκαμε πολλές φορές με το θέμα με τον κύριο Τσόλο και το αντιμετωπίσαμε το θέμα με τον κύριο Τσόλο και του ζητήσαμε δηλαδή Μα πρόκειται για εκτιμώντα. Μα βεβαίω πρόκειται για ένα εκτιμώντα που θέλει απλώ να επαναλάβει αυτό το οποίο είχαμε ζητήσει ήδη εμεί στον Επίτροπο για να παρέμβει πολύ πιο γρήγορα. Ο Μάρκ Ταραμπέλα. Πρόεδρε, εγώ ήθελα να πάρω το λόγο τώρα, διότι Σημερίζομαι μεν το νόημα της τροπολογίας Σιλβέστρης, αλλά λυπούμε για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται και κατατίθεται αυτή η τροπολογία. Δηλαδή, εδώ και τρεις μήνες έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες. Και εκφράζω τη θλίψη μου δηλαδή για τη διαδικασία. Το ελαιόλαδο είναι επίσης κάτι το οποίο μας καίει, αλλά η δυσκολία είναι σε όλους τους γεωργικούς τομείς, το βολιό κρέας, τα αυγά. Τέλος πάντων, εγώ σήμερα δεν θα αντιταχθώ στην προφορική τροπολογία. Άμα ψηφιστεί θα ψηφιστεί. Εγώ όμως θα καταψηφίσω για να εκφράσω την ε, διαμαρτυρία μου για τη διαδικασία. Δεν ξέρω, δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα για γαλακτοκομικό τομέα, α μιλήσουμε και για ελαιόλαδο, τότε γιατί να μην μιλήσουμε και για βόλιο κρέα. Λυπούμε δηλαδή, ενώ εδώ και τρει μήνες συζητάμε τι τροπολογίες, να κατατίθεται αυτή η τροπολογία μία ώρα πριν ψηφίσουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει η πολιτική μου ομάδα, μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει, αλλά εγώ θα καταψηφίσω. Ευχαριστώ Μάρκ. Σίγουρα δεν πρόκειται για την κλασική διαδικασία. Ο εισηγητή όμως τη λέει, ο Τζέιμ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Σιλβέστρη ε, που μας έκανε το απόγευμα λίγο πιο ενδιαφέρον από ότι ε, θα περνούσαμε διαφορετικά. Κοιτάξτε, εγώ ε, προτείνω να το δούμε θετικά. Ε, τον ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο πρότεινε την τροπολογία του, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν έχω πρόβλημα να ψηφίσουμε χωριστά σήμερα εδώ, αλλά να προσθέσω μια προϋπόθεση, μια ε, συνθήκη να το κοιτάξει το Κοινοβούλιο Υπηρεσίες ε, για να δούμε αν είναι παραδεκτή ή όχι η τροπολογία αυτή και αυτό που προτείνει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το ψηφίσουμε και να το υποστηρίξω, αλλά χρειάζεται έλεγχο. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι παραδεκτό. Γιατί υπήρξαν και άλλα θέματα που μπήκαν ε, ε, στην έκθεση και επειδή είναι νομοθετική, επειδή δεν ε, ήταν το αντικείμενο αυτό, το αφήσαμε απ' έξω. Ήταν εκτός τόπου και εκτός θέματος. Να το κοιτάξουν οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και μετά εγώ είμαι πρόθυμος να το δεχτώ. Αν μπορεί να συμφωνήσει ο κύριος Σιλβέστρης στη γενοδορία που δείχνω και εγώ και τη μεγαλοψυχία. να το υποστηρίξει κατά τμήματα ή χωριστή, συγγνώμη, χωριστή ψηφοφόρια. Ευχαριστώ, Τζιμ. Αν δεν υπάρχει επίσημη αντίρρηση στην προφορική τροπολογία θα ψηφίσουμε και μετά θα δούμε πώς θα ψηφίσουμε. Κανένας δεν είναι λοιπόν κατά. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία του κυρίου Σιλβέστρης και άλλων. Πέρας ψηφοφορίας. Περίμενε, περίμενε λέει ο πρόεδρος. Συγγνώμη. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία Σιλβέστρης. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ισοπαλία. Όχι, 19 ψήφισαν. Συγχαρητήρια κύριε Σιλβέστρης. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εγώ ήθελα επισήμω να υποσχεθώ κυρίω στον συνάδελφο Ταραμπέλα ότι δεν θα το ξανακάνω, δεν θα το ξανακάνω. Τελευταία φορά. Λοιπόν, συμβιβασμό γ, συμβιβασμό σε. Α, α, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, είχαμε και μερικέ άλλες τροπολογίες, Τι ξέχασα. Μία τροπολογία που δεν ψηφίσαμε, μου λέει η γραμματεία. Είναι η 43 Άλβες στη σελίδα 10. Ψηφίζουμε τη 43. Πέρας ψηφοφορίες. Τελειώνει η σελίδα, τελειώνει και η ψηφοφορία. 43. Ε, εγκρίνεται. Πάμε τώρα με τον συμβιβασμό Γ. Σε. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δέλτα. Συμβιβασμός Δ. Δέλτα. Ελληνικό. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Α, έχουμε την 57. Ψηφίζουμε ναι ή όχι, λέει ο πρόεδρος. Όχι, δεν ψηφίζουμε. Ωραία. Συμβιβασμός ε. Ψηφίζουμε πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός F λατινικό σίγμα τάφ ελληνικό. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβασμός G. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβασμός H. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβασμός Ι. Αρχίζει ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός J. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός K. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Την 93 Πατράων Εύες πρέπει να ψηφίσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 94 Ψηφίζουμε την 94, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός M, μη, πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 100, Ντελάνους μαγινές Αρχίζει η ψηφοφορία για, το συμβι... για την τροπολογία 100. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός όμικρον αλφα μικρό. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμό νη. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός όμικρον. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 112 τροπολογία. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός π. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Q. Συμβιβασμός Q. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τελικά συμβιβασμός R. Ψηφίζουμε. Συμβιβασμός R. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι, εγκρίνεται. Συμβιβασμός S. Ψηφίσατε όλοι για τον συμβιβασμό S. Εγκρίνεται. Νομοθετική πρόταση ούτως τροποποιημένη. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 31 υπέρ, καμία αποχή, 3 κατά. Ψηφίζουμε για το νομοθετικό ψήφισμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και στο τέλος τελική ψηφοφορία για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και δίνουμε εντολή στον εισηγητή μας για τη διαπραγμάτευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Μεγάλε James, συγχαρητήρια και κουράγιο. Όταν τα θέλει το λόγο, μης... για τον συμβιβασμό εσ. Μα δεν ψηφίσαμε την 11 του εισηγητή. Α, όχι, λάθος έκανα, ναι, ναι, ναι, λάθος έκανα, λέει ο κύριος Σταντά. Αγαπητοί φίλοι, ψηφίσαμε και το πακέτο για το γάλα. Το επόμενο ραντεβού είναι στις 7 το απόγευμα 4 Ιουλίου στο Στρασβούργο. Στρασβούργο λοιπόν, στις 7 το βράδυ στις 4 Ιουλίου. Τελείωσε η συνεδρία της Επιτροπής μας.